Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Πρόκειται για την ε, σύγκληση σε σώμα της Επιτροπής Προπολογισμών για την ε, θητεία 2014-2020. Έχω την τιμή να προεδρεύω ως απερχόμενος πρόεδρος της Επιτροπής αυτής Σας προτείνω να αρχίσουμε αμέσως γιατί έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Να ξέρετε ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες που χρειαζόμαστε, δεδομένες της σύνθεσης της Επιτροπής μας, δηλαδή υπάρχουν όλες οι γλώσσες πλην των Μαλτέζικων. Σε όλες τις συνεδριάσεις τη Επιτροπής μας να ξέρετε ότι θα υπάρχει αναμετάδοση στο διαδίκτυο μέσω webstream. Και να γνωρίζετε ότι μερικές φορές θα χρειαστεί και θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εάν λοιπόν, εάν λοιπόν υπάρχουν κάποιοι ευρωβουλευτές που δεν έχουν μαζί τους την κάρτα τους τότε όταν θα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, θα πρέπει να το λένε από την αρχή γιατί έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε προσωρινά μια νέα κάρτα όταν θα μπαίνετε στην αίθουσα. Λοιπόν, σήμερα για παράδειγμα, υπάρχει κανείς που να μην έχει την ηλεκτρονική του κάρτα μαζί. Γιάννους, είναι ένας νέος εδώ που ξέχασε φαίνεται σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι σκοπός της σημερινής μας συνεδρίασης είναι να συγκροτήσουμε το Προεδρείο πρώτα απ' όλα της Επιτροπής Προπολογισμών για την πεντετή αυτή. Θα κλέξουμε καταρχήν τον Πρόεδρο και στη συνέχεια θα κλέξουμε τέσσερις αντιπροέδρους σύμφωνα με το άρθρο 204 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς θα εκλέξουμε πρώτα τον Πρόεδρο και στη συνέχεια τους Αντιπροέδρους. διάφορα τακτικά μέλη έχουν ήδη ε, δώσει εξουσιοδότηση. Ο κύριος Παύλο Τζερόγκερόμπα πρώτα απ' όλα θα αντικαθαστήσει την κυρία Νεριάντα. Ο κύριος Τανιέλα Αγιώτα από το FTT αντικαθιστά τον κύριο Πέτερ Μάρκ. Ο κύριος Ντέρεκ Βόρθεν αντικαθιστά την κυρία Κλέρ Μούντι. Ο Κατή Περί από τους σοσιαλιστές αντικαθιστά τον κύριο Πολ Τάγκ. Υπάρχουν άλλες τέτοιες ε, αντικαταστάσεις, εξουσιοδοτήσεις. Όχι, καλώς. Συνεπώς, συνεχίζουμε. Πρώτο σημείο, εκλογή του πρέδρου. Εδώ χρειαζόμαστε απαρτία, ένα τέταρτο των μελών. Δέκα ευρωβουλευτές χρειάζονται. Είμαστε παραπάνω από 10. Προφανώς. Άρα έχουμε απαρτία. Ε, θέλατε το λόγο αγαπητέ συνάδελφε. Αντικαθιστώ. Επίσης ένα από τα μέλη της ομάδας ECR. Πρόεδρος, το σημειώνουμε. Ευχαριστούμε. Υποψηφιότητες. Υπάρχουν υποψηφιότητες στην Προεδρία. Κύριε Ζεράρ Ντεπρέ, πολύ χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ μεταξύ μας, μετά από λίγα χρόνια απουσία. Ντεπρέ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκω εδώ τους συναδέρφους. Εκ μέρους της ομάδας μου, με ιδιαίτερη χαρά προτείνω στην Προεδρία της Επιτροπής μας τον συνάδελφό μας Jean Artu. Ευχαριστούμε. Άλλη υποψηφιότητα παρακαλώ. Υπάρχει. Όχι από ό,τι βλέπω. Ζητώ από τον κύριο Ζων Αρτουή να μου πει κατά πόσο δέχεται να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής μας. Ναι, Πρόεδρε, δέχομαι. Ευχαριστούμε. Συνεπώς, διαπιστώνω ότι ο κύριος Ζων Αρτουή προτάθηκε από μια πολιτική ομάδα, από το Άλντε, σύμφωνα με τόσο προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 1 στο άρθρο 209. Διαπιστώνω ότι σύμφωνα με ε, το ίδιο σημείο στον κανονισμό αποδέχτηκε την πρόταση αυτή. Διαπιστώνω επίσης ότι βάση του άρθρου 204 σημείο 1 είναι τακτικό μέλος, πλήρες μέλος της Επιτροπής μας. Εξάλλου, έχει συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων βάσει του παραρτήματος αριθμός 1 του κανονισμού μας. Δεδομένου ότι είναι ο μόνος υποψήφιος για την Προεδρία, δηλώνω διαβοή ότι εκλέγεται στη θέση αυτή του Πρόεδρου. Jean Συγχαρητήρια και σας παραχωρώ την Προεδρία. Thank you, thank you, dear Thank you for your confidence. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Θα φροντίζω να ανταπεξέλθω στο έργο μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μόλις εκδηλώσατε στο πρόσωπό μου. Να γνωρίζετε ότι θα πράξω ό,τι είναι καλύτερο για να ανταποκριθώ στο έργο μου. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω τον Αλέν Λαμασούρ που προείδρευσε αυτής τη Επιτροπής με ιδιαίτερη ικανότητα που ε, στήριξε τον αγώνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήμασταν μέλη τη ίδια κυβερνήσεω, του κυβέρνηση του Αλέν Ζουπέ, ανάμεσα το 1995 και το 1997 όπου αυτός ως υπουργό ε, προπολογισμού και εγώ υπεύθυνο για την οικονομία και για την δημοσιοοικονομικά μπορώ να πω ότι είμαστε και ο ένας και ο άλλος ε, βασισμένοι στην ε, αυστηρότητα, στην ε, λιτότητα συγγνώμη, του προπολογισμού ή μάλλον στην ειλικρίνεια του προπολογισμού. Μέσα σε δύο χρόνια κατορθώσαμε να μειώσουμε από 6 σε 3% των το χρέος, ε, το, το έλλειμμα, συγγνώμη, του, προ, το δημόσιο έλλειμμα στη Γαλλία. Είναι γεγονός ότι χρειάστηκε να απολέσουμε, να χάσουμε τις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό είναι το τίμημα που χρειάστηκε να πληρώσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την εκλογή μου και για την επιλογή σας. Για να συμμετάσχω στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ξέρετε, η Επιτροπή Προπολογισμών είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα. Φυσικά το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολυετές και αφορά την περιοδο 2013 2014-2020. Σίγουρα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις και οι προκλήσεις δεν θα λείψουν. Καταρχήν διότι αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 2016 και ίσως ε, και νωρίτερα. Αυτή η αναθεώρηση είναι μια δημοκρατική απέτηση. Το κοινοβούλιο που μόλις εξελέγει θα πρέπει να πει τον γνώμη του πάνω στο πλαίσιο του ευρωπλισμού το οποίο θα αφορά το σύνολο της, ε, της ε, περίοδου θητείας. Χρειάζεται λοιπόν να προσέξουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αναθεώρηση όμως του, του δημοσιονομικού πλαισίου είναι μια αναγκαιότητα η οποία εμφανίζεται ευθύ εξ αρχή. Έχω υπόψη μου την ικανότητα απορρόφησης των υπολείπων προς εκαθάριση και τις νέες προτεραιότητες. Να υπενθυμίσω ότι τα υπόλοιπα προς εκαθάριση είναι η διαφορά ανάμεσα στις ε, δεσμεύσεις πληρωμών και της του πληρωμών και ανέρχονται σε πάνω από 220 δις, των οποίων τα 24 ε, δις είναι απαιτητά άμεσα. Νομίζω επίσης πως η ζώνη ευρώ θα μας απασχολήσει σε ό,τι φορά τη διακυβέρνησή της που οδηγεί στο να βρούμε ένα νέο προϋπολογισμό το μέσο δημοσιονομικής σταθερότητας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συνθήκης για τη Σταθερότητα, του Συντονισμού και τη Διακυβέρνηση, να βρούμε μια ικανοποιητική απάντηση, η οποία θα ικανοποιεί τις προσδοκίες των Εθνικών Κοινοβουλίων και τις χώρες της ζώνης Ευρώ και του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν είναι δυνατόν να ε, μας ικανοποιήσουν οι εξελίξεις μέχρι τούδε. Ε, <clears throat> θα πρέπει γενικότερα να σκεφτούμε το διοικητικό άχθος και τα δημόσια, δημόσια οικονομικά που θα μας ε, οδηγήσουν σε μια καλύτερη διαχείριση. Θα σας πρότεινα λοιπόν μια, ένα εγχείρημα προβληματισμού για να αντιμετωπίσουμε τον οδικό χάρτη. Και τις επόμενες ώρες πρόκειται να αποφανθούμε στις βασικές κατευθυντικές γραμμές του προορισμού 2015. Ευχαριστώ συνάδελφοι για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. So we have now to... Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στην εκλογή των αντιπροέδρων της Επιτροπής μας. Σας αναφέρω τα ονόματα των αναπληρωματικών που λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία. Είναι ε, αυτή που ανέφερε ο Αλέαν Λαμασούρ και αν υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή η αρμόδια πολιτική ομάδα πρέπει να μας πληροφορήσει. Υπάρχει κάποια αλλαγή? Όχι. Λοιπόν, το Πρέπει να αναφέρω ότι φυσικά υπάρχει απαρτία βάσει του άρθρου 208 του κανονισμού μας. Και ζητώ τώρα προτάσεις για τους αντιπρόεδρους. So, we have Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση για πρώτο αντιπρόεδρο. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποιος υποψήφιος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ του ΕΛΚ θα ήθελα να προτείνω για πρώτο αντιπρόεδρο τον Πέτρη Σαλβαμάρ. ο Πέτρης Αλβαμάρ. Ε, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα προς τον υποψήφιο, εάν συνενεί για την υποψηφιότητα αυτή. Βεβαίως, λέει, με μεγάλη χαρά. Ωραία. Οι προϋποθέσεις για, τον, για την εκλογή του εκπληρούνται. Έχει υποστηριχθεί από μια πολιτική ομάδα. δέχεται την υποψηφιότητά του, είναι πλήρως μέλος της Επιτροπής μας, έχει συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και είναι και ο μόνος υποψήφιος. Και προτείνω να τον κηρύξουμε εκλεγέντα διαβοής. Mr. Petri Would you... Σαλουαμάρα, ελάτε στα, προεδρικά θεωρία, παρακαλώ. Συγχαρητήρια. Thank Και ερχόμαστε τώρα στην εκλογή του Δευτέρου Αντιπρόεδρου. Έχουμε και εδώ την απαρτία. Έχουμε τώρα το δεύτερο αντιπρόεδρο, προτάσει για το δεύτερο αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Εξ ονόματο της Σοσιαλιστικής Ομάδος θέλω να προτείνω τον κύριο Γιάννη Γκάιερ για να είναι δεύτερο αντιπρόεδρο. Do you consent to be a candidate? Συμφωνείτε να γίνετε υποψήφιος, είστε υποψήφιος. Είστε πλήρως μέλος της ε, Επιτροπής μας, έχετε συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Υπάρχει κάποιος άλλος υποψήφιος. Όχι. Υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος λοιπόν για την θέση του δεύτερου αντιπροέδρου και σας προσκαλώ να τον εκλέξετε διαβοής. Congratulations, Jens Συγχαρητήρια. Ελάτε παρακαλώ στα προεδρικά θεωρία. Et maintenant l'élection du troisième. Ο τρίτος αντιπρόεδρος τώρα δεν είχα υπάρξει αλλαγή στους αναπληρωτές, υπάρχει πάντα η απαρτία και σας ζητώ υποψηφιότητες για τον τρίτο αντιπρόεδρο. Υπάρχει υποψήφιος για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του ΕΛΚ, προτείνουμε για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου τον Ζίγβερ Βάζιου Μούρεσαν. Δέχομαι την πρόταση αυτή. Μη υπάρχοντα άλλου υποψηφίου για τη θέση αυτή του τρίτου αντιπροέδρου και δεδομένου ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τα προαπαιτούμενα, ε, κηρύττω τον κύριο Ζίγκρετ Μουρεσάν, τρίτο αντιπρόεδρο και σας προσκαλώ να τον εκλέξετε διαβοήσου. Τον ίδιο να έρθει στα προεδρικά έδρανα. Ερχόμαστε στον τέταρτο αντιπρόεδρο. Δεν έχει υπάρξει αλλαγή στους αναπληρωτές, έχουμε πάντα απαρτία. Ζητώ υποψηφιότητες για τη θέση του τετάρτου ε, αντιπρόεδρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ του ΕΛΚ προτείνουμε για την αντιπροεδρία αυτή την Πατρίσια Σούλινγκ. Πατρίσια Σούλινγκ λέει ο πρόεδρος. Αποδέχεστε την υποψηφιότητά σας. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος Ευρώπης Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας θέλω να προτείνω τον κύριο Μαρκοζάνη. Μαρκοζάνη, μάλιστα. Κύριε Μαρκοζάνη, δέχεστε την υποψηφιότητά σας. Βεβαίως. Διαπιστώνω ότι έχουμε δύο υποψηφίους και οι δύο δέχονται να είναι υποψήφοι. Είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής μας και έχουν συμπληρώσει την δήλωσή τους για οικονομικά συμφέροντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω εξ ονόματος ομάδας μου των Πρασίνων να κάνω ένα σχόλιο για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν θεωρώ ότι είναι πρέπον οι μεγάλες ομάδες να αποφασίζουν να αποκλείσουν μια ομάδα από τις αντιπροεδρίες μόνο λόγω της προσωπικότητας του ηγέτη αυτής της ομάδας και του γεγονότος ότι κάποια μέλη αυτής της ομάδας είναι αντιτιθέμενα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό για μένα δεν είναι επαρκής λόγος για να αποκλειστεί η ομάδα από τα αξιώματα του Κοινοβουλίου. Διαφωνούμε βέβαια με την πολιτική θέση της ομάδας αυτής, αλλά υποστηρίζω την ανάγκη να πάρουν το EFD την τέταρτη αυτή αντιπροεδρία. Διαπιστώνω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο υποψήφοι. Θα πρέπει να ψηφίσουμε με μυστική ψηφοφορία. Και προτείνω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζω ότι ο καθένας σας έχει μία ψήφο. Πρέπει να βάλετε την ηλεκτρονική σας κάρτα στην ε, εσοχή, στο μηχάνημα. Η ομάδα του ΕΛΚ διαθέτει συνολικά 12 ψήφους. Οι σοσιαλιστές 11 το ECR 3, το ALDE 4, η πράσινη 3, το EFDD 3, και μία γεγραμμένη 3. πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων ο υποψήφιος. Αυτές θα είναι οι ψήφοι υπέρ. Οι αποχές δεν μετράνε. Ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες σας. Όσοι δεν έχουν τις κάρτες τους, τους δώσαμε νομίζω άλλες προσωρινές. Σωστά. Λοιπόν, επενθυμίσω τα ονόματα των υποψηφίων. Πρώτος υποψήφιος. Η κυρία Σούλιν. Της ομάδας των Πρασίνων, λέει ο πρόεδρος. Λάθος, συγγνώμη. Από τα ΕΛΚ είναι η κυρία Σούλιν. Ο κύριος Ζάνη είναι από το FDD. Λοιπόν, η κυρία Σούλιν είναι η πρώτη υποψήφια. υποψήφιο αριθμό 2 είναι ο κύριος Ζάνη. Αν ψηφίσετε για τον πρώτο, ψηφίζετε το πράσινο κουμπί για την κυρία Σούλινγκ και για τον κύριο Τσάνη ψηφίζετε αν πατήσετε το κόκκινο κουμπί. Θα ψηφίσουμε τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορία. Είδω το αποτέλεσμα. Ψήφισαν 31 ευρωβουλευτές. Είχαμε μία λευκή ψήφο. Συνεπώς 30 εκπεφρασμένες ψήφους. Η απόλυτη πλειοψηφία είναι 16 ψήφοι. Η κυρία Σούλινγκ είχε 20 ψήφους ο κύριος Ιωζάνη 10. Συνεπώς η κυρία Σούλινγκ εκλέγεται στη θέση του τέταρτου αντιπρόεδρου. Εκλέγεται συνεπώς η κυρία Σούλινγκ. Παρακαλώ να έρθετε κι εσείς εδώ στο Προεδρείο. Ε, signor Presidente, vorrei fare una Πρόεδρε, μια σύντομη δήλωση ως πολιτική ομάδα και ως Ιταλική Ευρωσοπία, κρίνουμε ότι τα όσα συνέβησαν αποτελούν σοβαρή παραβίαση, παραβίαση της δημοκρατικής αρχής διότι υπενθυμίζω πως θεμελιώδης αρχή που θα έπρεπε να βασίζεται ε, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, και της Επιτροπής μας ε, παραβιάστηκαν νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε ε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ευχαριστώ και τη μειοψηφία. Καταγράφω την δήλωσή σας. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρέμβαση. Πρώτα απ' όλα για να συγχαρώ τον πρόεδρό μας και τους άλλους αντιπροέδρους, τους αντιπροέδρους μας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Η επιτυχία σας θα είναι και δική μας επιτυχία. Έχουμε πολλές προκλήσεις που ανέφερε ήδη ο πρόεδρός μας και τις οποίες συμμεριζόμαστε. Υπάρχει βέβαια το θέμα των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό που μας απασχολεί είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της. Είναι προτεραιότητα για όλους μας η αύξηση της απασχόλησης. Συγχαρητήρια λοιπόν και είμαι σίγουρος ότι θα βρεθείτε, θα αρθείτε στο ύψος των ε, προκλήσεων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στον απερχόμενο πρόεδρο, τον Αλέν Λαμασούρ, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος, έθεσε την εμπειρογνωμοσύνη και την ικανότητά του στην υπηρεσία της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου μας. Θέλω λοιπόν να πω μερσή αλλά λαμασού για το εξαιρετό έργο σου. <clears throat> Και επίσης και για το αποτέλεσμα της ε, ε απόφασης που ελήφθη. Επεκράτησε η δημοκρατία, έγινε μια ψηφοφορία και οι ψήφοι της πλειοψηφίας είναι και αυτές ψήφοι σεβασμού προς τη δημοκρατία. Αυτό λοιπόν έλαβε χώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η λειτουργία της δημοκρατίας και θέλω λοιπόν να εκφράσω και την ευαρέσκειά μου για το αποτέλεσμα που επετεύθη με πλειοψηφία, με απόλυτη διαφάνεια, απόλυτο σεβασμό των κανόνων που διέπουν αυτή την εκλογή. Ευχαριστώ. Εντάξει, λοιπόν έχει περατωθεί η συγκρότηση του Προεδρείου μας και απλώς πρέπει να επιβεβαιώσουμε το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για το υπόλοιπο του 2014. Έχετε ενώπιον σας το χρονοδιάγραμμα αυτό. Και έχω και κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω. Η νέα Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει ένα σημαντικό ποσοστό νέων μελών. Γι' αυτό η Γραμματεία θα σας διανύμει ένα αριθμό εγγράφων, μεταξύ των οποίων το λεγόμενο Welcome Pack, τον απολογισμό των δραστηριοτήτων 2009-2014 και άλλες σχετικές πληροφορίες σε σχέση με τις ενεξελίξει διαδικασίες και ιδίως για τον προϋπολογισμό του 2015 και τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών για το 2014. <clears throat> Η πρώτη συνάντηση των συντονιστών για, ε, για κατεπήγοντα διορισμό εισηγητών, ιδίως για το Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης και για την ακρόαση του Επιτρόπου Γιάσεκ Ντόμινικ και την προετοιμασία του Τριλόγου θα λάβει χώρα στις 9.30 το πρωί την 10η ε, Ιουλίου πριν από τον Τρίλογο. Τα κόμματα θα πρέπει να δώσουν τα ονόματα των συντονιστών του στη γραμματεία το ταχύτερο δυνατό. Για το τριγωνικό διάλογο για τον προϋπολογισμό του 2015 οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τους εισηγητές του το ταχύτερο δυνατό. Από την κυρία Μπάλ, ε, θα, η κυρία Γκουαρδέα Σαουάλ θα επικυρωθεί ως Γενικός Εισηγητής για το 2015 και ο κύριος Γκαρίγκα ως εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2015 των άλλων θεσμικών οργάνων εκτός της Κομισιόν και αυτό θα, θα τον ε, αντικαταστήσουμε και επίσης και την κυρία Γιάνσεν ως, ε, ως υπεύθυνη για τον προπολογισμό του 2015 και επίσης για την κυρία Χολμάερ, η οποία είναι η αρμόδια για τον προπολογισμό 2014 για τα άλλα θεσμικά όργανα. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο στις 14 Ιουλίου στις 6.30 το βράδυ για μια μίνι ακρόαση του Ιασικ Ντάνατσεκ του υποψηφίου επιτρόπου. Η επόμενη τακτική μας συνεδρία θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στι 23 όλη τη μέρα. Η γραμματεία θα είναι σε επαφή σας για να καθορίσει το γλωσσικό προφίλ της Επιτροπής, το οποίο ε, στη συνέχεια θα εφαρμόζεται στις ε, τακτικές συνεδριάσεις. Κηρύττω τη λήξη της συνεδρίασης. Καλό τα μέλη της Επιτροπής και το προσωπικό να αποχωρήσουν διότι επίκειται μία άλλη συνεδρίαση στην ίδια αυτή αίθουσα. Σας ευχαριστώ.